Συνάδελφοι, όπω σα έλεγα, φτάσαμε στο σημείο 25 τη ημερήσια διάταξη τη Επιτροπή Διεθνού ανάπτυξη. Έχουμε από κοινού συνεδρίαση με την Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου, ΙΝΤΑ. Σα το έλεγα και χτε, αυτή την εβδομάδα θα ασχοληθούμε με διάφορα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι εβδομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προετοιμαζόμενοι για την 10η Δεκεμβρίου, την επέτειο της, παγκόσμ... της των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θα συζητήσουμε σήμερα για το... τη συμφωνία του ΟΗΕ για τις διεθνικές επιχειρήσεις και άλλες ε, επιχειρήσεις και την... το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα μας ενημερώσει η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για το πού βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις ε, επί της συνθήκης αυτής. Γνωρίζουμε ότι από το 2014 έχουν ξεκινήσει σχετικές διαπραγματεύσεις. Έχει ξεκινήσει μια ανοιχτή διακυβερνητική ομάδα, στόχος της οποίας είναι να καταλήξει σε μια διεθνή, ε, νομικά δεσμευτική συνθήκη, η οποία θα ρυθμίζει ε, την ευθύνη των διεθνικών επιχειρήσεων ε, και άλλων επιχειρήσεων να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το ερώτημα είναι Πώ παρευρέθηκε και τι ποιο ήταν το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Το ζήτημα είναι πολύ σημαντικό. Είχαμε εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισμα στι 4 Οκτωβρίου του 2018 με το οποίο ζητούσαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα κράτη-μέλη της να εμπλακεί με τρόπο υποκοδημητικό σε αυτέ τι διαπραγματεύσει του ΟΗΕ Προσπαθώντα να καταλήξουμε τελικά σε μια τέτοια νομικά δεσμευτική συνθήκη. Γνωρίζουμε Ποιε είναι οι θέσει των κρατών μελών. Νομίζω με μεγάλο ενδιαφέρον θα ακούσουμε την ενημέρωση από την κυρία Λουίσα Ράγκα, την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, είναι υπεύθυνη του Τμήματος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Θα δώσω το λόγο και στον κύριο Λάγκε. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά από έναν καθαρά εμπορική θεώρηση. Έχουμε να κάνουμε με λογοδοσία, με δέους επιμέλεια, που αποτελούν ένα πολύ βασικό κομμάτι του παιχνιδιού. Έχουμε τον κανονισμό για το ρηκτά από περιοχές με σειράξει. Ήταν πολύ σημαντικό βήμα αυτό. Η οδηγία για την υποβολή εκθέσεων, μη δημοσιονομικών εκθέσεων. Όσον αφορά την κατάσταση, είναι πολύ σημαντικό να εστιάσουμε σε αυτό το σημείο, το κομμάτι του εμπορίου και όχι μόνο ε, σε περιφερειακές ε, συμφωνίες. Να δούμε λοιπόν ποιες είναι οι εξελίξεις. Ο λόγος στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε να σας μιλήσουμε για αυτό το σημαντικό θέμα. Ε, για την υποστήριξη επίσης να σας ευχαριστήσουμε στην κοινή φωνή που έχουμε στα ανθρώπινα δικαιώματα. Συζήτησαμε ήδη το θέμα της δυναμικά της συνθήκης στην Ολομέλεια του Οκτωβρίου. Δεν θα επαναλάβω αυτά που ήδη υπόθηκαν. Ε, Στι 15 Οκτωβρίου έγινε η τελευταία συνεδρίαση στη Γενέβη της διακυβερνητικής ομάδας ε, υπήρξε μια κοινή συμφωνία για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα ότι το βασικό, ο βασικός προβληματισμός για το σχέδιο της συνθήκης ήταν την που είχαμε μια προτινόμενη συνθήκη και γι' αυτό το λόγο υπήρξε ε, επιφύλαξη. Σε γενικές γραμμές η αξιολόγηση της διαχείρισης του κύκλου αυτού συζητήσεων ήταν θετική σε σχέση με προηγούμενες συνεδριάσεις υπήρξε μια σχετική ουδετερότητα. Υπάρχουν όμως ακόμα ανησυχίε όσον αφορά και τη διαδικασία αλλά και το περιεχόμενο. Όσον αφορά το περιεχόμενο, το πρωτοδυνόμενο νομοθετικό με μέσο δεν καλύπτει όλες τις επιχειρήσεις, αφορά μόνο τις διεθνικές δραστηριότητες και δεν βασίζεται εξ ολοκλήρου στα, στις δεσμευτικές αρχές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δεν υπάρχει αναφορά στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών καν. Δεν υπάρχουν διορθωτικά μέτρα και δεν υπάρχει ευθυγράμμιση επομένως με τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ. Ζητήσαμε μία με ρόλο την προσέγγιση να υπάρξει διαφάνεια, προβλεψιμότητα και να βασίζεται η διαδικασία σε ε, ήδη υπάρχουσες πρακτικές ε, που ισχύουν για διακυβερνητικές ε, ομάδες. Το ψήφισμα πάνω στο οποίο βασίζεται θα πρέπει να ανανεωθεί. Αυτό δεν έγινε στην τελευταία ε, Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πολλές χώρες συμφωνούν με την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό θέλουμε να δούμε αν αντικατοπτρίζονται οι ανησυχίες μας στο αναθεωρημένο κείμενο που θα είναι διαθέσιμο τον Ιούνιο του 2019. Επιπροσθέτως, κάτι που επίσης συζητήθηκε με το Κοινοβούλιο είναι ότι δεν υπάρχει ε, ενδιαφέρον από πολλές χώρες για τη διαδικασία ε, όπως είπα, ο Καναδά, η Νορβηγία και άλλε χώρε οι οποίε δεν συμμετέχουν ε, στις ε, συνεδριάσεις, μόνο 27 χώρες από αυτές που παρευρέθηκαν έλαβαν το λόγο ε, σε μια εβδομάδα συζητήσεων. Αξιολογούμε παράλληλα τα αποτέλεσμα της τέταρτης συνεδρίασης και την πιθανότητα αυτή η διαδικασία να οδηγήσει σε μεγαλύτερη προστασία για τα θύματα και επίση να υπάρχει ισότιμη ε, μεταχείριση έναντι των επιχειρήσεων. Το συζητάμε αυτό με τα κράτη-μέλη, με την κοινωνία των πολιτών, με τις επιχειρήσεις. Και ανυπομονούμε να δούμε και ποια είναι η δική σας η άποψη και για το περιεχόμενο αλλά και για τη διαδικασία. Θα ήθελα να προσθέσω ότι αναφορικά με τη διαδικασία αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεγάλο ιστορικό στην εφαρμογή ε, νομοθεσία ε, που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, επίση σε, σε προγράμματα δράσης και επίσης να ε, πολλές επιχειρήσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζουν από μόνε τους ήδη τις αρχές αυτές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Υπάρχουν ήδη ε, άλλες ε, οδηγίες και κανονισμοί πάνω στους οποίους μπορούμε να βασιστούμε, πώς είναι αυτή της εταιρική ευθύνη, ε, της, ε, ο κανονισμός για το ρηκτά που περιέχει με σειράξει και Θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση σε διορθωτικά μέτρα, να υπάρχει να υπάρχουν ισότιμες ευκαιρίες και να τηρηθούν τα διεθνή στάνταρ. Αυτό αυτή είναι η δική μου δήλωση και είμαι διαθέσιμη να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση. Um, Σας ευχαριστούμε. πρώτος, παρακαλώ. Ή πρώτη μάλλον. Ευχαριστώ πολύ, Λίντα. Μιλώ εξ ονόματός μου αλλά και εξ ονόματος ενός συναδέλφου του Μάκη Λάντερ που δεν μπορεί να είναι παρόν, Ροντρίγκε Περέρο, γιατί ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βλέπουμε ότι ε, υπάρχει μια γενικότερη υποστήριξη από όλε τι πολιτικέ ομάδε. Αυτό φάνηκε και στο ψήφισμα το οποίο εγκρίναμε στις 4 Οκτωβρίου. Η ΕΜΑ μαζί με άλλου ευρωβουλευτέ από άλλε πολιτικέ ομάδε ξεκίνησαν μια εκστρατεία κοινοβουλευτική προκειμένου οι ε, βουλευτέ σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο να δημιουργήσουν μια σφαιρική καμπάνια πίσω από τη δεσμευτική αυτή συνθήκη, την προτινόμενη. Γιατί ουσιαστικά αναγνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να λειτουργούμε με τον τρόπο που λειτουργούμε τώρα. Χρειαζόμαστε ένα πλήρες πλαίσιο προκειμένου να μπορούμε να εντάξουμε σε αυτό όλες τις διαφορετικές διατάξεις που υπάρχουν από τον ένα τομέα στον άλλον, από τη μία περιοχή του κόσμου στην άλλη, για να έχουμε ένα σφαιρικό τελικά εργαλείο και θεωρώ ότι εδώ οι κατευθύνες γραμμές των εθνών είναι χρήσιμες αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν επαρκούν από μόνε του. Γιατί αν αρκούσαν οι εθελούσιε πρωτοβουλίε, τότε θα ζούσαμε σε έναν ιδανικό κόσμο όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα θα προστατεύονταν παντού. Βλέπουμε συχνά όμω ότι οι εθελούσιε αυτέ πρωτοβουλίε δεν αρκούν. Γι' αυτό το λόγο, ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για την υλοτομία, την ξυλία, για τα ορυκτά τα οποία προέρχονται από εμπόλεμε ζώνε, ζητήσαμε δεσμευτική δέουσα επιμέλεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να βγούμε από το αδιέξοδο αυτό στο οποίο βρισκόμαστε, όπου μας λένε ότι υπάρχει πρόβλημα με τη διαδικασία, πρόβλημα με το περιεχόμενο. Μπορούμε και τα δύο αυτά να τα συζητήσουμε, και θα δείτε ότι υπάρχει μια γενική υποστήριξη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το πεδίο εφαρμογή που θα πρέπει να έχει αυτό το δεσμευτικό εργαλείο, για το τι θα πρέπει να περιέχεται στο εργαλείο αυτό και το καθεξή. Ακριβώ όμω επειδή βρισκόμαστε τώρα σε ένα αδιέξοδο, ακριβώ επειδή δεν έχουμε εγκρίνει μια συγκεκριμένη εντολή ω Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε μια διοργανική συζήτηση για το τι θα πρέπει να γίνει στα πλαίσια των ΗΕ. Και η προσωπική μου άποψη είναι ότι ε, αυτό προκαλεί ιδιαίτερη αγανάκτηση στου ευρωβουλευτέ και σε μένα, γιατί ξέρουμε ότι εξελίσσεται η συζήτηση. Υπάρχουν πολλέ χώρε ανά τον κόσμο που τοποθετούνται αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένα κείμενο από το οποίο εμεί θα μπορούσαμε να πούμε τι μας αρέσει και τι όχι ή βάσει του οποίου θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε συμμαχίε με άλλε χώρε. Θα ήθελα λοιπόν πέρα από όλα αυτά να μου πείτε ποια είναι η άποψή σας όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή, μπορούμε να συμβάλλουμε κάποια χρονική στιγμή και εμεί διαπραγματεύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πότε θα γίνει αυτό. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι φτάνουμε πλέον στο τέλος της περίοδου εκείνη όπου καλούμεθα απλώ να είμαστε σιωπηλοί παρατηρητέ, χωρί να έχουμε μια ξεκάθαρη εντολή ω Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει περάσει οκτώ ολόκληρα ψηφίσματα και δύο ψηφίσματα έχουν να προέρχονται από την Συνέλευση Ευρωπαϊκή Ένωση Λατινική Αμερική. Γνωρίζουμε λοιπόν το ζήτημα, ξέρουμε τι θέλουμε να πετύχουμε για τα επόμενα στάδια. Και μια τελευταία παρατήρηση. Αυτό που καθιστά την κατάσταση αφόρητη πραγματικά είναι ότι βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή έχουν καταβληθεί τόσες πολλές προσπάθειες, τόσοι πολλοί πόροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς επίσης και από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για τις διαπραγματεύσεις αυτές. Έχουν καταβληθεί φοβερές προσπάθειες να προσελκύσουμε χώρες εταίρους για να καταφέρουμε να πείσουμε 20 χώρε να μπουν στι διαπραγματεύσει αυτές, γιατί πραγματικά δεν θα πρέπει να είναι μόνο οι πιο πλούσιε και δυνατές χώρε που θα συμμετέχουν στη διαπραγμάτευση τη συνθήκη αυτή. Προσπαθούμε πραγματικά να προωθήσουμε πάρα πολύ το ζήτημα αυτό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των διεθνικών επιχειρήσεων αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούν να συμμετέχουν και οι χώρες εκείνες, οι πολίτες εκείνοι, οι πολίτες λέω, οι οποίοι έχουν ζημιωθεί πραγματικά από τη δράση κάποιων διεθνικών επιχειρήσεων που δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό για μένα είναι απαράδεκτο. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προωθούμε τα δικαιώματα για τους πολίτες και τους κανόνες για τις επιχειρήσεις. Και δεν το κάνουμε αυτό, δεν θα καταφέρουμε ποτέ να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στην ε, ευρωπαϊκή, στο ευρωπαϊκό εμπόριο και στη διεθνή δράση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Μπέρντ Λάνκ έχει, έχει το λόγο. Ένα σημαντικό λόγο στην κατάσταση στα κράτη-μέλη και ίσω θα πρέπει να αναλογιστούμε λίγο παραπάνω ποιο είναι το σκεπτικό των κρατών μελών ποια είναι η συμμετοχή των κρατών μελών στην ε, Γενέβη και πώς θα συνεχίσουμε τη διαδικασία ώστε να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για το ποιος ε, συμμετέχει, που δίνεται έμφαση και τι κάνει το κάθε κράτος μέλος. Ε, Μαρία Αρένα. Μαρία Ρένα. Ευχαριστώ. Υποστηρίζω πλήρως αυτά που είπε η συνάδελφο Τζουντ. Έχω ένα ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποια ήταν εκείνα που υποστήριξαν ουσιαστικά μια νομικά δεσμευτική διεθνή συνθήκη. Ποτά δεν το μάθαμε αυτό. Μήπως μπορείτε να μας το πείτε σήμερα. Ποιοι ήταν εκείνοι που σας υποστήριξαν αυτό που είπε η Jude είναι ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχει μια υποστήριξη από όλες τις πολιτικές ομάδες, το οποίο δεν φάνηκε μόνο στο ψήφισμα, αλλά οποτεδήποτε είχαμε μια ψηφοφορία για την ε, υποχρεωτικό χαρακτήρα που πρέπει να έχει ιδέουσα επιμέλεια. Εμείς πάντοτε υποστηρίζουμε αυτή την προσέγγιση την υποχρεωτική. Λέτε ότι θα θέλατε να ξέρετε ποια είναι η θέση του Κοινοβουλίου. Η θέση του Κοινοβουλίου είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη ακόμα και όταν η πρόταση η οποία μας υποβάλλεται προβλέπει εθελοντικό χαρακτήρα, το μετατρέπουμε ή προσπαθούμε στον τριμερή διάλογο να τη μετατρέψουμε σε υποχρεωτική. Αυτή είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να μας ενημερώσετε για το ποια είναι η θέση των κρατών μελών. Θα ήταν χρήσιμο για να μπορέσουμε και εμείς να αναλάβουμε εκστρατείες πολιτικές, έτσι ώστε να δούμε τελικά ποιοι είναι εκείνοι που θέλουν να υπερασπιστούν τα δικαιώματα των πολιτών και ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι ε, προτιμούν μια εθελοντική προσέγγιση. Σα ευχαριστούμε κυρία Λόλα Σάντσες. Ευχαριστώ Λίντα. το ιστορικό αυτής της σχέση τη Ευρωπαϊκή Ένωσης με την επιβολή κανόνων στις επιχειρήσεις είναι ε, τεράστια και έχει και διφορούμενη. Εγώ το θυμάμαι εδώ και χρόνια. Αυτή τη φορά έχουμε υποστηρίξει ένα ψήφισμα στις 4 Οκτωβρίου, πάρα πολύ σημαντικό, αλλά βρισκόμαστε εκεί που βρισκόμαστε πριν από ένα χρόνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα, τα θύματα μάλλον αυτές της, ε, αυτών των προβλημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παντού στον κόσμο περιμένουν από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει το σθένος που πρέπει και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να διαφοροποιηθούμε από τις θέσεις που παίρνει η κυβέρνηση Τραμπ και οι Ηνωμένε Πολιτείες. στη Γενέβη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δυνατότητα να πιέσει έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια νομικά δεσμευτική συνθήκη για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις επιχειρήσεις. Αυτό καλή το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο περιλαμβάνει και πολύ συγκεκριμένε προτάσει για τα θέματα τα οποία θα έπρεπε να θέσει στο τραπέζι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω πέρασε καιρό, πέρασαν εβδομάδε και δεν ακούσαμε ούτε μία πρωτοβουλία να ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλά πράγματα μπορούν να βελτιωθούν. Πολλά πράγματα μπορούν να βελτιωθούν, για παράδειγμα, σε σχέση με τη διαδικασία. Όμω θεωρώ ότι είναι θλιβερό το θέμα που παρακολουθούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Γενέβη, το μόνο που να προσπαθεί να κάνει είναι να φρενάρει αυτού που προσπαθούν να σταματήσουν τη συνθήκη, αντί εμεί να έχουμε πιο φιλόδοξου στόχου του οποίου να επιδιώκουμε, πιο φιλόδοξου από αυτού που μα παρουσιάζουν. Για παράδειγμα, να γίνεται ξεκάθαρο στη συνθήκη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα υπερτερούν οποιασδήποτε άλλη υποχρέωση. Αυτό είναι απαραίτητο. Δεν είναι καινούργια αυτά που σα λέω. Όλα αυτά βρίσκονται στο ψήφισμα τη 4 η Οκτωβρίου. Όταν βλέπω τι ρόλο έπαιξε η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Γενέβη, δεν βλέπω μια Ευρωπαϊκή Ένωση την οποία μπορώ να υποστηρίξω και την οποία πιστεύω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει, είχε και πρέπει να συνεχίσει να έχει τα ανθρώπινα δικαιώματα ως σημαία της. Δεν μπορούμε να μιλούμε για εθελοντικό χαρακτήρα. Ε, ήδη πολλοί πολίτες έχουν γυρίσει την πλάτη τους σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ρωτώ, λοιπόν, πώς θα συνεχίσετε να, παρα, να παρευρίσκεστε να συμμετέχετε στην Γενέβη. Θα προσπαθήσετε να αξιοποιήσετε το γεγονός ότι είμαστε ένα σημαντική κομπλόκ ε, κρατών ε, ή απλώς θα προσπαθείτε να ε, κάνετε μια διαχείριση των συνεπειών της, της, των θέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Σας ευχαριστώ. Θα ζητήσω από τους συναδέλφους να μην μακρηγορούν, γιατί δεν θα έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Κυρία Χάιτι Χάουταλα, έχει ζητήσει το λόγο. Κύριος... Κυρία Μίμερ και ο κύριος Σάρλ ε, Γκέρενς. Γρήγορα σας παρακαλώ, κυρία Χάουτελα. Θα ήθελα να γνωρίζω περισσότερα πράγματα όσον αφορά τα σημεία από την οποία διαφωνεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με αυτό το σχέδιο συνθήκης και να δούμε τελικά αν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ασκήσει επιρροή για να αλλάξει τα πράγματα αυτά τα οποία βαίνουν κακώς και κυρίως όσον αφορά το πεδίο της εφαρμογής και συμφωνώ ότι δεν θα πρέπει αυτό το οποίο αποφασίζουμε να ισχύει μόνο για τις διεθνικές εταιρείε, αλλά για όλες τις εταιρείε. γιατί ε, το προφίλ των επιχειρήσεων αλλάζει, η παγκόσμια λυσίδα εφοδιασμού αλλάζει, θα πρέπει να καλύπτονται λοιπόν όσο δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις. Μήπως ε, θα ακουστεί πιο ηχηρά η φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν στις διεθνείς αυτές διαπραγματεύσεις ε, μπορούσε να αρχίσει να εφαρμόζει και αυτή καλύτερα τι κατευθύνες γραμμέ των Ηνωμένων Εθνών. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καν ένα ευρωπαϊκό σχέδιο όσον αφορά τι επιχειρήσει και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σα ευχαριστούμε κυρία Μίνε και μετά ο Σαρλ Γκέρεν. Θα είμαι πολύ σύντομη. Δεν έχουμε διερμηνία στα Ολλανδικά, έτσι δεν είναι. επομένω, θα χρειαστεί να μεταφράσω λίγο γρήγορα το κείμενο αυτό που έχω μπροστά μου, το οποίο είναι στα Ολλανδικά. Αυτή τη στιγμή συζητάμε για ένα δεσμευτικό εργαλείο για την ε, προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο των επιχειρήσεων. Σας συγγνώμη, δυσκολεύομαι, λέει η ομιλήτρια. Είμαι πολύ ικανοποιημένη με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ήλπιζα πραγματικά ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση θα χρησιμοποιούσε περισσότερο το ψήφισμα αυτό στην δική τη την τοποθέτηση. Ο λόγο για τον οποίο η συνθήκη αυτή είναι πολύ σημαντική είναι διότι οι διεθνικές αυτές εταιρείες δεν ακολουθούν το εθνικό δίκαιο. Και αυτό βέβαια αποτελεί άμεση επίπτωση της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, όπου οι πολυεθνικές κάνουν οτιδήποτε μπορούν προκειμένου να μην ακολουθούν και να μην δεσμεύονται από το εθνικό δίκαιο. Και έχουμε πολλές επιχειρήσεις οι οποίες καρφίζονται οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε προκειμένου να μην είναι υπόλογε για τις χειρότερες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα αρνητικό το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία στο ζήτημα αυτό, το αποδυναμώνει τελικά, επικεντρωνόμενοι κυρίως στις εθνικές εταιρείες. Μα καταλαβαίνετε ότι το πιο σημαντικό σημείο τη συνθήκη αυτή και ο λόγο για τον οποίο πρέπει να έχουμε μια διεθνική, μια συγγνώμη, δεσμευτικά συνθήκη είναι ακριβώ για να καλύψουμε και τι διεθνικέ εταιρείε. Υπάρχουν διάφορε εθνικέ πρωτοβουλίε, οι οποίε θα, έπρεπε να είχαν προβληθεί περισσότερο από τι εθνικέ αντιπροσωπείες που συμμετέχουν σε πραγματεύσει Γενέφη. Θα μπορούσατε να μιλήσει και Ολλανδικά, λέει η πρόεδρο τελικά, ο Σάγλ πολύ γρήγορα. Ολοκληρώνουμε μέσα σε τέσσερα λεπτά, λέει Πρόεδρο. Συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπε η Μαρία Ρενά. Ιδίω ε, όσον αφορά την ε, απαράδεκτη, αξιολύπητη πραγματικά στάση των κρατών μελών. Μα τα κράτη-μέλη τελικά είναι ο ασθενή κρίκος τη Ευρωπαϊκή ε, Ένωση αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι σε μια εποχή που ο Τραμπ προσπαθεί να καταλύσει όλα τα συστήματα διεθνού συνεργασία, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αντιτάξει το παράστημά τη για να τα προασπίσει. Και απευθυνόμενο και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, πρέπει να σα πω ότι όλη αυτή η συζήτηση είχε γίνει και στα πλαίσια του ΟΣΑ. Υπάρχουν και εκεί κατευθυντήρε γραμμέ, από τον ΟΣΑ δηλαδή. Θα ήθελα να γνωρίζω λοιπόν τι γίνεται με τις συζητήσει και τι διαπραγματεύσει στα πλαίσια του ΟΣΑ, όπου συμμετέχουν οι πιο πλούσιες και εκβιομηχανισμένες χώρες. Νομίζω λοιπόν ότι και εκεί πέρα το ζήτημα θα μπορούσε να έχει καλυφθεί πλήρω. Ευχαριστούμε πολύ η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράσης. Θα προσπαθήσω να απαντήσω. Συμφωνώ πλήρως ότι είμαστε προθλητές στα ανθρώπινα δικαιώματα. Θέλουμε να παραμείνουμε, αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Γιατί δεν, ε, ε, γιατί δεν συμμετείχαμε στη διαδικασία, το κάναμε τις προηγουμένες φορές, αλλά όχι πλήρως και το θέμα ήταν ότι δεν είχαμε την εντολή να το πράξουμε αυτό. Χωρίς εντολή δεν μπορεί να διαπραγματευτείς. Επίσης οι ανησυχίες σας είναι γνωστές, τις έχω επαναλάβει γιατί δεν θέλουμε να εστιάσουμε μόνο σε διεθνικές δραστηριότητες αλλά και σε εγχώριες δραστηριότητες είναι για να δημιουργήσουμε ισότιμε ευκαιρίες. Αν δεν καλύψουμε ένα κομμάτι των επιχειρήσεων τότε δεν υπάρχει ισότητα ή σε αντιμετώπιση. Όσον αφορά τη θέση των κρατών μελών, τα κράτη μέλη ε, είναι, ε, έχουμε τη γεμοφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. θα έπρεπε να παρέμβουμε στην αρχή και να είμαστε ξεκάθαροι ως προς το ποιες είναι οι θέσεις μας, τι πράττουμε και τι προσδοκούμε από αυτή τη διαδικασία. Τα κάτι υποστήριξαν αυτή τη θέση και υπήρξε μια ενιαία Ευρωπαϊκή Φωνή τελικά. Όταν ρώτησα ποια είναι η αξιολόγηση του Ευρωκοινοβουλίου και να ακούσω τις απόψεις δεν είχε να κάνει με το ψήφισμα της 4ης Οκτωβρίου. Φυσικά και το διάβασα και το εκτιμώ. Η ερώτηση μου ήταν ε, ότι τώρα που έχει ολοκληρωθεί η συνεδρίαση και κάποια κράτη-μέλη ήταν ε, παρόντα στη διαδικασία, αν είδανε πρόοδο ή δεν είδαν πρόοδο, τι θα κάνουμε στη συνέχεια, το ημερολόγιο, Λοιπόν, προς το παρόν, η Πρόεδρος ε, λέει ότι οι διερμηνείς μπορούν να αποχωρήσουν και ότι η να θα συνεχιστεί στα αγγλικά